La Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Ξαναρχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Τα πρακτικά για την χθεσινή συνεδρίαση έχουν διανεμηθεί. Το επόμενο θέμα είναι η κοινή συζήτηση για την Τραπεζική Ένωση και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Πρόκειται για την εισήγηση Tyson και την εισήγηση Giggold. Και δίνω τον λόγο για τέσσερα λεπτά στην κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί Επίτροπε, νομίζω